Λοιπόν, ξεκινήστε ψάχνοντας πρώτα απ' όλα τις κάρτες, τις κάρτες ψηφοφορίας, γιατί θα αρχίσουμε να ψηφίζουμε τον, κατερχήν το σχέδιο προϋπολογισμού. Είναι η ώρα. Δεν περιμένω. Να περιμένω λίγο. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Καθίστε με τις κάρτες ψηφοφορίας. Θέλω να καλωσορίσω όλους τους ε, νεοαφιχθέντες. Ήδη χαιρέτησα τμήμα των ε, βουλευτών, τους διερμηνείς ε, και τους υπαλλήλους που ήταν παρόντες στην προηγούμενη συνεδρίαση. Εύχομαι αυτή η νέα σχολική χρονιά, λέει η Πρόεδρος, να είναι παραγωγική. Πρώτο, Έχουμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη και αν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη αλλά ο κύριος Αδόψε έχει κάτι να πει. Η κυρία Άδοψη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω. Προτού όμως υιοθετήσουμε την ημερήσια διάταξη, θα ήθελα να παρακαλέσω να προβλέψουμε στα διάφορα να συζητηθεί η όλο και πιο σοβαρή κατάσταση σχετικά ε, με ε, το γάβρο με το Σαφρίδι ε, το Βόρειο Ατλαντικό, με συγχωρείτε, και νομίζω ότι η Επιτροπή αυτή θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να το συζητήσει, διότι η κατάσταση ε, γίνεται όλο και πιο δύσκολη στην περιοχή την οποία εκπροσωπώ και θα ήθελα να συμφωνήσει όλοι οι ομίγυροι στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ κυρία Ντότς. Este tema, que es de gran interés para todos, pero sobre todo para un gran número de que su sector está afectado por una serie de Σας ευχαριστώ λοιπόν που θίξατε το θέμα. Εγώ ήδη το εξήγηλα στην ε, συνεδρίαση των συντονιστών ότι θα φύγατε σίγουρα το θέμα και θα το εξετάσουμε στο τέλος της ημερήσιας διάταξης. Προσθέτουμε αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη και η συνεδρίασή μας αναμεταδίδεται στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Πάμε στην έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 22ης ε, Ιουνίου και της 14ης και 15ης Ιουλίου του 2010. Έχετε τα έγγραφα στο φάκελό σας και αν δεν έχετε, αντι... δεν έχετε αντιρρήσεις θα εγκριθούν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ανακοινώσεις Προέδρου δεν έχω τίποτα να πω. Πάμε στο πέμπτο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έκθεση της γνωμοδότησης της κυρίας Ρόντουστ σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2011 σχετικά με την Αλία. Κυρία Ρόντουστ, θέλετε να πείτε κάτι, μπορούμε να ψηφίσουμε κατευθείαν. Ψηφίζουμε κατευθείαν. Θα ψηφίσουμε πρώτα τις τροπολογίες δημοσιονομικού χαρακτήρα και μετά τις τροπολογίες επί της γνωμοδότησης. Πρώτον, θα ψηφίσουμε την 6723. Θα σας λέω τον αριθμό της τροπολογίας. 6723 της κυρίας Φράγκα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ένας πράσινος παραπάνω. Δύο. Εγώ δεν ξέρω αν το μηχάνημα έχει πάντα δίκιο, αλλά ας ξαναψηφίσουμε. Λοιπόν, ξαναψηφίζουμε για την 6723. Πάλι ένας πράσινος παραπανήσιος. Πέρασε κανείς τους πρασίνους και δεν το πήραμε χαμπάρι. Μα ποιοι πράσινοι είστε εδώ. Συντονίστρια μπορείτε να μου το ξεκαθαρίσετε λίγο το θέμα. Εγώ είμαι και ο κύριος Μπεσέτα από τους Πρασίνους. Ο, δεν υπάρχει κανείς άλλος από ό,τι βλέπω. Ο κύριος Χάνσον και ο κύριος Ρωμέβα δεν είναι εδώ. Γι' αυτό και εγώ είπα, μα κανείς ε, προσιλητήσατε κανέναν ε, στο δόγμα σας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και δεν το πήρα χαμπάρι. Τέλο πάντων, δεν ξέρω μπορεί να συνέβη σε κανέναν άλλον. Εμένα δεν μου συνέβη. Τέλο πάντων, λοιπόν, ωραία, εντάξει, ψηφίζουμε. Πέρα ψηφοφορία. Τώρα Πράσινος παραπανήσιος δεν ξέρω ποιος. 15-3 λοιπόν εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 67-08 και την 6732 μαζί που είναι ίδιες τις εισηγήτριες. Λοιπόν, αρχίζουμε την ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Ψηφίζουμε την 6709 και την 6736 της εισηγήτριας που επίσης είναι ίδιες. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται ομόφωνα. Ψηφίζουμε τις ε, τροπολογίες 6710 και 6733 της εισηγήτριας που επίσης είναι ίδιες. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνονται ομόφωνα. Ψηφίζουμε την 6711 και την 6738 που επίσης είναι ίδιες. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα πάλι δύο ίδιες ε, τροπολογίες, την 6712 και την 6739 της εισηγήτριας. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες. Δεν κρίνεται. Ψηφίζουμε την 6701 του κυρίου Φερέιρα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 6713 της κυρίας Φράγκα. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 6702 του κυρίου Φεραίρα. Αρχίζει ψηφοφορία. izquierda. Απορρίπτεται. Λοιπόν, τώρα θα ψηφίσουμε ένα σχέδιο πιλότο. Είναι η τροπολογία 6705 του κυρίου Φερέιρα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δύο ταυτόσιμες τροπολογίες, 67-14 και 67-26 της εισηγήτριας. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες. Εγκρίνεται ομόφωνα. Ψηφίζουμε. Πάλι δύο ταυτόσιμες τροπολογίες, την 67-15 και την 6727 της εισηγήτριας και αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες. Εγκρίνεται ομόφωνα. 6716 και 6728 της εισηγήτριας πάλι ταυτόσιμες αρχίζει η ψηφοφορία. <coughs> Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Ψηφίζουμε άλλες δύο ταυτόσιμες τροπολογίες, την 6717, την 6729 της εισηγήτριας, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Ψηφίζουμε τις 6718 και 6730 της εισηγήτριας. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνω ομόφωνα. Ψηφίζουμε την 6706, τροπολογία για ένα σχέδιο πιλότου του κυρίου Φερέρα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. «6703 του κυρίου Φερέρα, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Έγκρινεται 10 υπέρ, 8 κατά και 2 αποχές. Ψηφίζουμε για τη γραμμή 110702 που έχουμε τρεις τροπολογίες. Η πιο διαφοροποιημένη είναι η 6704 του κυρίου Φερέρα. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε λοιπόν τις επόμενες τροπολογίες, στην 67, 19, 67, 31 για την ίδια γραμμή του προϋπολογισμού είναι ταυτόσιμες, η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. λοιπόν, έχουμε την τροπολογία 6740 αφορά σε δύο γραμμές του προϋπολογισμού. Η κυρία Λούεβιν είναι η εισηγήτρια και, και ζητά ξεχωριστή ψηφοφορία. Ε, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θα ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα μείωση 4 εκατομμυρίων ευρώ για τη γραμμή 110801 αρχίζει ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίες απορρίπτεται και ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα αύξηση κατά 4 εκατομμύρια ευρώ της γραμμης 11.08.05.02 που αφορά στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ελέγχου. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 11 και δύο αποχές. Ψηφίζουμε την 6720 και την 6734 για την 110801 που είναι επίσης ταυτόσιμες και που θέλουν να αποκαταστήσουν το ποσό του σχεδίου προϋπολογισμού. Αρχής ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. Ομόφωνα. Ψηφίζουμε τις δύο τροπολογίες μαζί, την 6721 και την 6735 της εισηγήτρες. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Ομόφωνα. Ψηφίζουμε πάλι δύο ταυτόσιμες τροπολογίες, 6722 και 6737 της εισηγήτριας. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ζούμε στη συνέχεια την 6707 του κυρίου Φερέρα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε μία τροπολογία για ένα σχέδιο πιλότου, είναι η 6700 του κυρίου Φερέιρα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 67-24 για ένα σχέδιο πιλότο της εισηγήτριας. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 11 ψήφους υπέρ και 9 κατά. Έχουμε την τροπολογία 67-25 της συγκήτρες για άλλο ένα σχέδιο πιλότο, αρχής ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 15 υπέρ, 2 ε, κατά. Τώρα ψηφίζουμε τη γνωμοδότηση στο σύνολό της. Ψηφίζουμε την τροπολογία της κυρίας Ρόντους. Πέρας ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τον συμβιβασμό 1 της εισηγήτριας. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 17-2 Καταπίπτουν. Ψηφίζουμε την πέντε της κυρίας Φράγα, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τέσσερα της κυρίας Ρέιμερς. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Έξι του κυρίου Γκαρίγα Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. απορρίπτεται 12-6 Τρία του κυρίου Καντέκ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 της κυρίας Φράγκα καταπίπτει μπαίνει στο συμβιβασμό 1, το ίδιο και η 8 της κυρίας Ρέιμερς και η εννέα του κυρίου Γκαρίγα Πογέδο. Ψηφίζουμε λοιπόν τώρα δύο ταυτόσημες ε, τροπολογίες, τη 10 και τη 11. Η πρώτη είναι της εισηγήτριας, αρχίζει. Όχι. Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, καταπίπτει αν περάσει ο συμβιβασμός ένα. Συγγνώμη λοιπόν. 12 λοιπόν του κυρίου Καντέκα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Λοιπόν, 13 συμβατεί με τη 14. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 14 του κυρίου Φερέιρα, αρχίζει ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Λοιπόν, Ρέιμερς 15, αρχίζει ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 16 του κυρίου Στίβενσον. Συμβατή. Με την 15. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 17 της κυρίας Λουεβίν. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τον συμβιβασμό 2 της εισηγήτριας. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν η 18 της κυρίας Ρέιμερς, η 20 του κυρίου Καντέκ και η 19 της κυρίας Φράγκα, 21 Φερέιρα λοιπόν. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 6. Ο κύριος ε, Καντέκ που είναι ο συντάκτης της τροπολογίας 22 μας έστειλε μήνυμα ότι αποσύρει την τροπολογία του. Ψηφίζουμε και υποστηρίζει τον συμβιβασμό 3. Λοιπόν ψηφίζουμε τον συμβιβασμό 3 και αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Καταπίπτει η τροπολογία Σάντσος Πρεσέδο, 24 της κυρίας Φράγα. Ψηφίζουμε 25 του κυρίου Καντάκ. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 26 της εισηγήτριας. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα 27 της κυρίας Ρόντους. Θα αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 28 της εισηγήτριας. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 29 της εισηγήτριας. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 30 της εισηγήτριας. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Ψηφίζουμε συνολικά λοιπόν την πρόταση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 18 υπέρ. Κανένας κατά, δύο αποχές. Συγχαρητήρια κυρία ρόντους και σα συγχαίρω για όλη την συμβιβαστική προσπάθεια που κάνατε για να πετύχουμε δηλαδή και την πλειοψηφία σε αυτό το σώμα. Σας ευχαριστώ ειλικρινά. Επόμενο σημείο Πω πω εμένα σήμερα μου πουλαχεί να δουλέψω διπλά λέει η Πρόεδρος. Λοιπόν, για τον κύριο Άμαν μπερδεύτηκα εδώ με την εισήγηση του κυρίου Γκάλαχερ, είπα το 7, εξήγηνα το 7 πριν από το 6. Λοιπόν, πρόκειται για την τροποποίηση του κανονισμού 2187 2005 του Συμβουλίου που αφορά την απαγόρευση διαλογής αλευμάτων ανώτερης κατηγορίας και τους περιορισμούς αλίες ε, όσον αφορά τη χωματίδα και το καλκάνι στα ύδατα της Βαλτικής θάλασσας, των Μπέλτς και του Σάουντ. Η συγητής είναι ο κύριος Γκρόμπετσιν. Τον Ιούλιο μας είχε παρουσιάσει η Κομισιόν την πρώτη της θέση, να την ακούσουμε όμως και σήμερα. Να ακούσουμε μάλλον τον εισηγητή σήμερα για να μπορέσουμε δηλαδή 19 Σεπτεμβρίου να συζητήσουμε το θέμα. Κύριε εισηγητά έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι Έχουμε εδώ πέρα μια πρόταση έκθεσης ε, της Επιτροπής η οποία είναι τεχνικής ε, φύσεως και αφορά τους ε, περιορισμούς όσον αφορά την εποχή της αλληλείας, ειδικά για τη Χωματεία και το Παλκάνι. Στο σημείο 1 όμως αναφέρεται ένα πολύ σημαντικό θέμα, και αυτό είναι το να σταματήσει η πολιτική των απορρίψεων, η οποία πρακτική ακολουθείται ευρύτατα μέχρι σήμερα. Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι το πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να μας απασχολήσει όλους, ειδικά στα κράτη εκείνα μέλη τα οποία βρέχονται από την Βαλτική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τους ψαράδες γιατί το σύστημα βεβαίως των απορρίψεων ήταν πάρα πολύ επιβλαβές και η Κομισιόν και στο παρελθόν το είχε αμφισβητήσει πολλές φορές. Θα ήθελα όμως εδώ πέρα να επισημάνω κάτι συγκεκριμένο που συνδέεται με την εγκατάλειψη αυτής της ε, πρακτικής. Γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα, καθώς ε, μία πτυχή εδώ πέρα δεν ε, ταιριάζει, δεν είναι συμβατή με την ιδέα την ίδια της αηφόρου ε, αλληλείας και εδώ πέρα μιλάω για την αλληλεία βεβαίως της βιομηχανικής αλληλείας γιατί άλλο η βιομηχανική αλληλεία και άλλο η παραδοσιακή αλληλεία μικρής κλίμακας και βεβαίως ε, στην περίπτωση της βιομηχανικής αλληλείας θα πρέπει να απαγορευτούν οι ε, απορρίψεις οτιδήποτε πιάνετε θα πρέπει να καταγράφετε και να αποτελεί αντικείμενο εμπορία και να φτάνει βέβαια στην εκτήρια σχολά. Όμω υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ πέρα και το πρόβλημα αυτό αφορά την ε, αλληλεία σε βιομηχανική κλίμακα. Υπήρχε ο κανονισμός 2026 ο οποίος αναφέρει συγκεκριμένα πως η αλληλεία βιομηχανική κλίμακας δεν καλύπτεται από κανέναν ε, έλεγχο, ειδικά στην Βαλτική. Και γι' αυτό είναι τόσο σημαντική αυτή η τροπή Είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί είναι εξαντλημένα τα αποθέματα αυτή τη στιγμή, πάρα πολύ ειδικά αυτό της ε, Ρέγκας ε, στη Δυτική Βαλτική είναι εξελιμμένο. Οπότε αν δεν υπάρχει απολύτως κανένας έλεγχος η κατάσταση θα χειροτερέψει και άλλο. Και φτάνουμε λοιπόν στην πολιτική αυτή των απορρίψεων. Και εδώ πέρα βρίσκεται η πραγματική απειλή, ο πραγματικό κίνδυνο. Οπότε το ερώτημά μου προ την Κομισιόν είναι το εξή. Πώ προτείνει η Κομισιόν να προχωρήσουμε. Έχει κάποια ιδέα για την φύση του κινδύνου που παρουσιάζουν, παρουσιάζει η πολιτική των απορρίψεων στην βιομηχανική κλίμακα αλληλεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπα, και όσον αφορά και τον ε, μπακαλιάρο και το ψάρι αυτό το αλλιεύουν, ε, το υπεραλλιεύουν, ε, το πιάνουν στα 30 μέτρα και μετά το πετάνε. Η κατάσταση λοιπόν είναι σαφής. Πρέπει να σταματήσει αυτή η πρακτική, δεν, ε, δεν το συζητάμε. Τώρα λοιπόν φτάνουμε στο ζήτημα ε, και της χωματίδας και του καλκανιού. Και εδώ πέρα έχω κάποιες ε, αμφιβολίες για να είμαι ειλικρινής. Έκανα κάποιους υπολογισμού και φαίνεται πως μέρος μόνο της Βαλτικής καλύπτεται από τις ε, κλειστές αυτές σεζόν, όπως λένε. Η υπόλοιπη περιοχή είναι εκτός ε, του πεδίου εφαρμογής. Ανέλησα λοιπόν το ζήτημα και είδα τις περιοχές 25, 26 και 28 και εδώ πέρα οι ποσότητες οι οποίες αλλιεύονται φτάνουν τους 100 τόνους, οπότε είναι σχεδόν αμεληταίο. Δεν υπάρχει λόγος να μιλήσουμε για κλειστές σεζόν. Εκεί όμως έχουμε κλειστές σεζόν, ενώ σε άλλες ε, περιοχές όπως ε, στο Belts και στο Sound και σε άλλους τομείς έχουμε ποσότητες ε, εκατοντάδων χιλιάδων τόνων τα δεδομένα αυτά είναι της Eurostat που σας λέω και δεν έχουμε καμία κλειστή σεζόν. Γι' αυτό έχω τις αμφιβολίες μου και αυτό είναι το ερώτημα που απευθύνω προς την Κομισιόν. Τι σκοπεύει δηλαδή να κάνει. Τι θα γίνει με το πρόβλημα αυτό με την ε, κλειστή σεζόν. Τι θα γίνει με τις διαφορετικές περιοχές της Βαλτικής. Όπως θα πρέπει να θεωρήσουμε την ε, έννοια αυτή ολόκληρη των ε, κλειστών σεζόν. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω και την Κομισιόν, ε, ιδιαίτερα την κυρία Ελίζα Μπόργκες για την συνεργασία μας και ελπίζω έτσι να συνεχιστεί και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Eh, Κανείς δεν θέλει το λόγο. Η εκπρόσωπος της Κομισιόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Όσον ε, αφορά την ε, απαγόρευση αυτή σε σχέση με την βιομηχανική αλληλεία, εμείς θεωρούμε πως η βιομηχανική αλληλεία δεν έχει τεράστια επίπεδα απορρίψεων, ακριβώς λόγω της φύσης ε, της αλληλεία αυτής. Τα αλληλεύματα δεν διαχωρίζονται ε, μεταξύ για ανάλογα με το μήκος ή το είδος ε, συνήθως χρησιμοποιείται όλο το αλίευμα και εξάλλου αλλιεύεται μόνο ένα είδος. Ε, οπότε είναι μικρό το ποσοστό. Όμως ισχύει αυτό για κάθε αλία στην Βαλτική και προφανώς για την βιομηχανική αλία ισχύει η απαγόρευση αυτής της πρακτικής. Τώρα όσον αφορά τις κλειστές αυτές περιοχές, οι κλειστές περιοχές υπάρχουν και δημιουργήθηκαν πριν από λίγα χρόνια στον σχετικό κανονισμό του συνολικού αλλιεύματος και βέβαια στόχο έχουν να προστατεύσουν το γόνο του καλκανιού και όχι βεβαίως ε, για να πούμε ποια θα πρέπει να είναι η ψηλότερη ελίευση. Σύμφωνα λοιπόν με Αυτά τα οποία μας λένε οι επιστήμονε. δεν υπάρχει λόγος για να προστατεύσουμε το γόνο να αλλάξουν ούτε οι περιοχέ ούτε οι εποχέ. Βεβαίω, να υπενθυμίσω πω οποιαδήποτε αναθεώρηση θα απαιτήσει μια επιστημονική αξιολόγηση και αναθεώρηση των τεχνικών μέτρων της Βαλτικής, τα οποία βεβαίως θα παρατείνουν την αξιολόγηση αυτής της πρότασης και δεν θα τεθεί ενισχύ η απαγόρευση διαλογής. Ε, να σας πω λοιπόν πως εδώ πέρα μιλάμε απλά για μια αλλαγή διατάξεων που υπάρχουν όσον αφορά το, τη συνολική ποσόστοση του αλεύματος και δεν σκοπεύουμε να αναθεωρήσουμε αυτά τα μέτρα Απλά μιλάμε για αλλαγή των νομικών απαιτήσεων και να πάνε στον κανονισμό τεχνικών μέτρων. Ευχαριστώ. Κύριε Ισηγητά, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Κύριε Ρόντουστ. Ευχαριστώ. Τώρα ε, είμαι κάπως ενοχλημένη διότι βεβαίως αλλάζουν πάλι οι ποσότητες και βλέπουμε ότι υπάρχει υπερβολική υπεραλίευση και άλλωστε πρέπει να αντιμετωπίσουμε και μία νέα επιστημονική αξιολόγηση. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι αν τραβήξει αυτή η κατάσταση εμείς θα υποταγούμε. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά αλλιεύματα και ε, τα αποθέματα τα λιευτικά όλο και μειώνονται είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε στο μέλλον και εσείς ε, λέγετε ότι ε, η βιομηχανία έχει αξιοποιήσει όλα τα λιεύματα αλλά δεν το καταλαβαίνω διότι βλέπω ότι υπάρχουν ορισμένα λιεύματα που επιτρέπονται μόνο σε συγκεκριμένα αυτό δεν ισχύει για τη βιομηχανία. Τι γίνεται, ο καθένα κάνει ό,τι θέλει. Είμαι πολύ ενοχλημένη και θα ήθελα να έχω πιο ακριβεί εξηγήσει. παρακαλώ. Η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Όταν ε, ε, μίλησα ότι πετούν ε, τα ε, ψάρια που δεν επιθυμούν σύμφωνα με τις πληροφορίες μου σημαίνει ότι δεν αξιοποιούνται αυτά τα προβλήματα δηλαδή το και ε, ε, το θέμα αυτό ε, για τις απορρίσεις είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με τα την παρεπίπτοντα αλία και δεν είναι κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνεται ή στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απλούστατα αυτή τη στιγμή ε, δεν το αντιμετωπίζουμε και είναι ένα θέμα το οποίο θα εξετάσουμε στο μέλλον όσον αφορά την πολιτική μας αλλά υπάρχουν μέτρα τα οποία ούτως ή άλλως ε, λαμβάνουμε υπόψη και ε, υπάρχουν τεχνικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται και ε, θα αξιολογηθούν μέσα στα πλαίσια της ε, αναθεωρήσεως της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ευχαριστώ την Κομισιόν και τον εισηγητή. Να σας πω ότι στις 29 Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστεί η έκθεση και 5 Οκτωβρίου λίγη προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Τελειώσαμε με το 6, πάμε στο 7. Συμφωνία με τη Χιλή, ο κύριος Γκάλαχερ είναι εισηγητής και ζητούμε την σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Το συζητήσαμε το θέμα στην τελευταία συνεδρίαση, ο κύριος Γκάλαχερ δεν είναι εδώ γιατί ε, δεν μπορούσε να έρθει και μου ζήτησε να παρουσιάσω εγώ το θέμα. Και εγώ, που ξέρετε ποιο είναι το ενδιαφέρον μου για το θέμα, θα περιοριστώ στην γνωμοδότηση του κυρίου Γκάλαχερ. Αν μου κάνετε καμιά ερώτηση μετά, θα απαντήσω κατά συνείδηση. Ξέρετε λοιπόν ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο δημιουργεί εμπορικές συγκρούσεις. Δεν πρόκειται εδώ για περιβαλλοντικό πρόβλημα, αλλά για εμπορικό. Είχαμε ένα πρόβλημα στη δεκαετία του 90 με τη Χιλή που ο της ψάρευε σε διεθνή ύδατα χωρίς τις απαραίτητες άδειε, διότι η Χιλή ποτέ της δεν συμμετείχε και δεν θέλησε να συμμετάσχει σε διεθνείς οργανισμούς. Τώρα βέβαια έχει προχωρήσει σε κάποια διαβήματα, αλλά μέχρι τώρα δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, μία ισπανική οργάνωση Λοιπόν, ε, οι Ισπανοί αλλοίς ε, μετράτες ε, είπαν ότι υπάρχει μία παραβίαση του άρθρου 5 της Συμφωνίας στα πλαίσια για το θέμα φόρτωσης-εκφόρτωσης και επίσης ένα πρόβλημα με το άρθρο 11 που, που δημιουργούσε εμπόδια στην εισαγωγή ξηφία στην Χιλή. Θεωρήθηκε λοιπόν ότι η Χιλή έθετε φραγμούς σε αυτού του τύπου την αλία και κατέθεσε μια καταγγελία στην ΠΟΕ, ο αρμόδιος επίτροπος. Το 2001 είχαμε μια προσέγγιση μεταξύ Χιλής και Ευρωπαϊκής Ένωσης για να λυθεί αυτή η σύγκρουση. Διακόψαμε την προσφυγή στην ΠΟΕ, την διακόψαμε, δεν την αποσύραμε, την αναστήλαμε απλώς για να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία μεταξύ Χιλής και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η προσωρινή συμφωνία που λειτουργήσε από το 2001 και μετά, λειτουργήσε πάρα πολύ άσχημα. Και όπως λέει και ο εισηγητής, έφυξε όλο το στόλο αλίας ξηφία, που αλλιεύει σε διεθνή ύδατα, όχι μόνο στη Χιλή, αλλά και στο στόλο ανοιχτής θάλασσας, που επίσης ψαρεύει στα ίδια διεθνή ύδατα και που αντιμετωπίζει προβλήματα εκφόρτωσης. Δηλαδή, αντί να λυθεί το πρόβλημα, επεκτάθηκε το πρόβλημα και σε άλλους στόλους, όχι μόνο δηλαδή το στόλο αλίας του Ξηφία, αλλά και του στόλους ανοιχτής θάλασσας. Η εσωτερική χιλιανή νομοθεσία δημιούργησε συνεχώς μεγαλύτερα προβλήματα τόσο στο θέμα της αλλίας του, ψυχή, ψηφία όσο και στο στόλο ανοιχτού πελάγους. Εγώ δεν αμφισβητώ καθόλου μα καθόλου ούτε την καλή θέληση της Κομισιόν ούτε την καλή θέληση των χιλιανών. Το 2008 ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις και κατέληξαν σε κάτι το αντίστοιχο με την προσωρινή συμφωνία η οποία δεν λειτουργήσε ποτέ. Οπότε η... ο κλάδος που πλήττεται από αυτή τη συμφωνία κατέθεσε προσφυγή λέγοντας ότι πρόκειται για την ίδια συμφωνία με την προηγούμενη. Αλλά η Κομισιόν μας λέει ότι εδώ πρόκειται περί διεθνούς δικαίου. Αλλά άμα πρόκειται περί διεθνούς δικαίου δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί εδώ χρειάζεται ειδική συμφωνία με τη Χιλή. Με το θέμα δηλαδή των λιμανιών και της εκφόρτωσης κλπ. Και υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα το οποίο αναφέρει ο εισηγητής και το ανακάλυψε τον Αύγουστο σε κάτι συζητήσεις που είχε με τον, με τον σχετικό επίτροπο. Η Κομισιόν είχε πει και έχω εδώ τα κείμενα ότι δεν θα αποσυρθεί ποτέ η καταγγελία. Έχει ανασταλεί. Αλλά Η καταγγελία υφίσταται. Και ότι θα αποσυρώταν άμα λυνόταν το πρόβλημα. Εμεί την ανακαλύψαμε όμως, ότι ακόμη έχει αποσυρθεί η καταγγελία πριν υπογραφεί η συμφωνία. Αλλά και η Ισπανική κυβέρνηση το αγνοούσε πλήρως το θέμα. Και αντιβαίνει απόλυτα με τις υποσχέσεις της Κομισιόν. Δεν θα φλιαρίσω άλλο. Ξέρετε ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν χρειάζεται πολλές φλιαρίες. Ο κύριος Γκάλαχερ λοιπόν συστήνει να καταψηφίσουμε. Διότι εγώ τώρα μιλάω εξ ονόματος του εισηγητού αλλά και όλη της Επιτροπής αισθανθήκαμε ότι όλη η Επιτροπή ότι μας δουλεύουνε διότι μας είχαν υποσχεθεί κάτι και κάναν ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν, εγώ λέω, είπα αυτά τα οποία ήθελε ο εισηγητής να πω και θα δώσω το λόγο στον κύριο Σάντσες Πρεσέδο. Εγώ θέλω να σταθώ στην έκθεση Γκάλαχερ. Δεν θα μιλήσω σε άλλα, για άλλα θέματα. Πρόκειται για, μια, για ένα πρόβλημα, για μια σύγκρουση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Χιλής. Πρόκειται για κάτι που ξεκίνησε στα τέλη του 1998, είχαμε μια καταγγελία της ΝΑΠΑ και από το 2001 και μετά υπάρχει και μία προσωρινή συμφωνία για την αναστολή, που προβλέπει την αναστολή της διαδικασίας δηλαδή, και η ΠΟΕ πολλές φορές επανέλαβε τις ε, δυσκολίες <coughs> και εγκρίναμε ένα νέο πλαίσιο 2008, από το 2008 και μετά ένα νέο πλαίσιο για να προχωρήσουμε. Εγώ θεωρώ όμως ότι το πλαίσιο το οποίο τίθεται σήμερα κάνει ένα βήμα, άρα πρόκειται για ένα θετικό πλαίσιο. Δημιουργεί ένα καλύτερο κλίμα. Πρόκειται για μια χώρα με την οποία έχουμε συμφωνίες, συνεργασίες, δεν πρόκειται για κάτι παράλογο. Θεωρώ λοιπόν ότι η έκθεση είναι αρκετά κακόπιστη διότι εκφράζει δυσπιστία προς ε, τον εταίρο. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε κάνει βήματα μέχρι σήμερα για να μπορέσουμε να έχουμε έναν διαπιστωμένο έλεγχο και από τις δύο πλευρές. Η Χιλή θέλει να περιφρουρήσει τον οικονομικό της χώρο. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση τη θέλει να διατηρήσει την αλλιευτική της ικανότητα σε διεθνή ύδατα. Να σταθώ εγώ σε μερικά συγκεκριμένα σημεία Λέμε εδώ <coughs> ότι η χιλή στερείται πολυμερούσα διάστασης. Ότι δεν έχει καθόλου συστήματα. Μιλάμε εδώ για το θέμα επίσης το ραντάρ, για τη διαπίστωση των πλοίων κλπ. Ορίζεται μία αναφορά στην διαμετακόμιση και μεταφορά θα έχουμε και τρία νέα λιμάνια για την εκφόρτωση. Και τίθεται και ένα σύστημα ε, νέο. Εμείς με τη Χιλή έχουμε μία συμφωνία συνεργασίας. Πρέπει λοιπόν να διαμορφώσουμε μία κουλτούρα συνεργασίας. Το status quo δεν σημαίνει ότι είναι η καλύτερη κατάσταση. Σημαίνει ότι η κατάσταση τελματώνει. Το σημαντικό για μας είναι να εξελιξόμεθα. Και εδώ έχουμε σαφείς βελτιώσεις. Εγώ τώρα δεν έχω καμία πληροφορία σχετικά με αυτά που μας είπε η πρόεδρος για την ΓΑΤ, λέει ο μιλητής εννοώντας την ΠΟΕ. Και το θέμα δηλαδή της απόσυρσης της προσφυγής. Και εδώ αυτό το οποίο λέγεται στην έκθεση ότι η αιτία του προβλήματος είναι οξυφίας και άλλα συγκεκριμένα είδη, ε, όχι, δεν βρίσκεται εκεί το πρόβλημα, είναι ένα καθαρό, καθαρά μεθοδολογικό πρόβλημα, πρέπει να λυθούν όλα τα προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να βρεθούν λύσεις. Εμείς πιστεύω ότι με αυτή τη συμφωνία τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει ε, προόδους. Θα έλεγα λοιπόν να υπερψηφίσουμε τη συμφωνία. Δεν έχω κανένα άλλο εναλλακτικό κείμενο που να μου λέει ποια θα είναι η καλύτερη λύση. Κοιτάστε, για μένα η καλύτερη λύση, λέει η Πρόεδρος είναι μια καλύτερη διαπραγμάτευση της συμφωνία. Λοιπόν, επαναδιαπραγμάτευση. Η Κομισιόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που δίνετε την ευκαιρία στην Επιτροπή να επανέλθει στο θέμα αυτό επί του οποίου έχει ήδη εκφραστεί. Θα ήθελα να περιοριστώ σε τρεις σύντομες παρατηρήσεις για να μην επεκτείνω χωρίς λόγο τη συζήτηση. Υπάρχουν πολλά στοιχεία στην έκθεση αυτή με την οποία συμφωνούμε. Διότι όπως είπατε κυρία Πρόεδρε, η συνεργασία είναι μια δύσκολη ιστορία η οποία χειροτέρεψε με μια εμπορική εμπλοκή. Δεν πρέπει όμως να κοιτάμε μόνο το παρελθόν αλλά και μπροστά. Για πρώτη φορά η Χιλή προτείνει με αυτή τη διμερή συμφωνία μία σειρά από εγγυήσει και δεσμεύσεις. Είναι λοιπόν ε, ενδιαφέρον για τους Ευρωπαίους να τις αξιοποιήσουν και να προχωρήσουν. Στην έκθεση του κυρίου Γκάλαχερ λέγεται ότι η καλή πίστη των χιλιάνων ε, ούτως ή άλλως διακυδεύεται. Οπότε ε, δεν μπορούμε έχουμε ε, εκ να αποφύγουμε ε, κάθε ε, συμφωνία με τη Χιλή που είναι βασικό εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο λόγω των προβλημάτων του παρελθόντος. Πρέπει να ε, γνωρίζουμε και να θυμόμαστε τι συνέβη αλλά να προχωρήσουμε και η κατάσταση είναι σημαντική για τους Ευρωπαίους γι' αυτό και διμερώς προτείνονται διάφορες λύσεις, διάφορες ο οπισθοχωρείς από πλευράς της Χιλής που είναι προς όφελός μας, που είναι ε, προς όφελος Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Λοιπόν, ε, βέβαια ίσως δεν είναι η ιδεώδη συμφωνία την οποία θα επιθυμούσαμε, αλλά σε διεθνείς ε, συζητήσεις δεν υπάρχουν τέτοιες ιδεώδεις λύσεις. Δεύτερον, θα ήθελα να ενημερώσω το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη σχετικά με την απόσυρση της περιπτώσεως από τον ΠΟΕ. Όλοι ενημερώθηκαν για την απόσυρση αυτή ε, του περιπτώσεως από τον ΠΟΕ. Τώρα όμως υπάρχει μία παρανόηση διότι ε, χρησιμοποιήθηκε η συνήθις οδός για την απόσυρση από τον ΠΟΕ όπου οι εμπορικοί εταίροι ασχολήθηκαν ε, στα πλαίσια του ΠΟΕ δηλαδή στα πλαίσια της της Επιτροπής ασχοληθήκαμε εμείς ε, στα πλαίσια του Συμβουλίου η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και οι συνδικαλιστές. Ίσως όλοι λοιπόν δεν έχουν ακολουθηθεί οι απόλυτα σωστές διαδικασίες αλλά σεβαστήκαμε όλους τους μηχανισμούς και δεν υπάρχει καμία επιθυμία εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραβλέψει τον βασικό ρόλο ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό. Το τρίτο θέμα που θα ήθελα να σημειώσω είναι τα συμφέροντα των Ευρωπαίων γιατί η έκθεση Γκάλαχερ λέγει ότι εδώ δεν ικανοποιούνται οι τράτες των Ισπανών αλλά στις τελευταίες επαφές που είχαμε με τους εμπλεκομένους ήταν ότι τους ενδιέφερε πολύ αυτή η ρύθμιση ίσως λοιπόν έχουμε χωριστή αξιολόγηση θα προσπαθήσουμε να τους ενημερώσουμε αλλά αυτές είναι οι πληροφορίες που διαθέτουμε. Μπορούμε να το συζητήσουμε εκτός συνεδριάσεως, αλλά αυτά τα στοιχεία έχουμε και πιστεύουμε ότι οι Ευρωπαίοι συγκεκριμένα αλλά και οι τράτες της Ισπανίας ειδικώ πρέπει να δεχθούν αυτά που μας προτείνει τώρα η Χιλή διότι εάν δεν τα δεχθούμε στο μέλλον θα είμαστε σε πολύ πιο αδύναμη θέση για να έχουμε καλύτερα εχέγγυα. Οπότε είτε τώρα τσεπώνουμε αυτά τα τα οποία μας δίδονται ή επειδή υποψιαζόμαστε τους χιλιάνους να μην είναι ειλικρινείς πλήρως γιατί αύριο θα αλλάξουμε γνώμη επ' αυτού. Και αν αυτό σκεφτόμαστε ουσιαστικά, γιατί τόσα χρόνια διαπραγματευόμαστε με τους χιλιάνους. Εάν πιστεύουμε κατά βάθο ότι δεν, δεν είναι ειλικρινείς οι χιλιάνοι, σταματήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Πράγμα το οποίο δεν είναι ε, ε, δεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντική εταίρη μας, έχουμε πολλές συναλλαγές, το βλέπουμε με τις διμερείς συμφωνίες για τον Ξηφία. Βλέπουμε επίσης ότι για πρώτη φορά η Χιλή συμμετέχει εις την οργάνωση της Αλίας στο Νότιο Ατλαντικό οπότε ε, μπορεί να μην έχουμε όλες τις λύσεις αλλά πρέπει να κοιτάξουμε να αποκομίσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε σήμερα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να ηρεμήσω και να απαντήσω. Εγώ πιστεύω ότι η Επιτροπή έχει μια διασπορά αρμοδιοτήτων και είναι πολλοί οι επίτροποι που ασχολούνται με το ίδιο θέμα. Ξέρω ότι για πολλούς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μετράει καθόλου. Και 14 Ιουλίου το συζήτησε εδώ το Κοινοβούλιο και ακούσαμε τι είπε η αρμόδια επίτροπος. Τώρα εσείς μπορεί να χάνετε τα αυγά και τα πασχάλια, δηλαδή εσείς ε, που ασχολείστε με το εμπόριο να μην ξέρετε τι κάνουν αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με, με, με, με την αλία. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι εδώ υπάρχει σύγχυση. Εσείς είπατε ο κλάδος συμφωνεί. Εγώ μίλησα με τον κλάδο στις 27 Αυγούστου και μου είπε ο κλάδος διαφωνούμε ριζικά. Εντάξει, ο λόγος σας ε, κατά του δικού μου. Κάπου λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα. Κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνουμε. Εσείς λέτε ή θα δεχθούμε αυτό ή τίποτα. Μα εσείς ε, πιστεύετε ότι η Χιλή κάθε φορά πρέπει να μας καπελώνει και να αποδεχόμαστε εμείς όπως έγινε και στην προηγούμενη συμφωνία αυτό που η Χιλή θέλει για τη Χιλή αυτή ήταν μια πρωταρχική συμφωνία. Ποτέ δεν θα είχε υπογράψει η Χιλή τότε άμα είχαμε θέση. Εγώ τότε ήμουν ε, υπουργό στην Ισπανία. Η Χιλή κάθε φορά μας επιβάλλει το τι πρέπει να κάνουμε. Αν λοιπόν αυτό είναι διεθνές δίκαιο τότε ας πληρωθεί το, κοινο, το διεθνές δίκαιο. Και υπάρχει αυτή η προσωρινή συμφωνία 2001-2008 διότι δεν χρησιμεύσε σε τίποτα. Και όχι γιατί λόγω κακής θέλησης της ισπανικής κυβέρνησης, αλλά λόγω κακής θέλησης της Χιλή. Διότι ποτέ δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν τα πλοία. Παρά τη συμφωνία. Και κάθε φορά τα ίδια. Και τα ίδια. Οι χιλιανοί δεν θέλουν ποτέ να δεχθούν μαθήματα από τους άλλους. Θέλουν να επιβάλλουν σε όλους την εφαρμογή του χιλιανού νόμου. Και άμα δεν, το δέχ, δεν δέχεται το χιλιανό νόμο, κανένας δεν μπορεί να εκφορτώσει. Και όλα αυτά, όσες φορές γίνανε καταγγελίες στην πόλη, δεν πέρασαν ποτέ Δείτε τι έγινε και με την Αυστραλία. Εσείς τι κάνατε, αποσύρατε τώρα την καταγγελία που δεν έπρεπε να κάνετε και δεν κάνετε τίποτα. Τίποτα πια στα χέρια μας, το διεθνές δίκαιο, το οποίο όμως επαφίεται στο τι θα της καπνίσει τη χιλής να κάνει. Λοιπόν, ας διαπραγματευτούμε ένα νέο μνημόνιο τόσο με τη συμμετοχή των ε, ψαράδων ξηφία και του στόλου ανοιχτής θάλασσας που είναι οι ενδιαφερόμενοι. Η λύση για μένα λοιπόν είναι να διαπραγματευτούμε μία νέα συμφωνία. Αυτή είναι η θέση μου. Η λέει να το απορρίψουμε απλώς. Ο κύριος Σάντσες Πρεσέδο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συμφωνήσω με δύο πράγματα που αναφέρθηκαν. Πρώτα, με την πρόταση απόφασης. Να αποσυρθεί η συμφωνία μετά από την έγκριση. Αλλά εδώ όμω θα έπρεπε να είναι συνεπής η Κομισιόν και να τα κάνει αυτά τα οποία λέει. Αλλά ε, εγώ θέλω να σας πω επίσης και κάτι άλλο, ότι ο κλάδος ανησυχεί σημαντικά. Όμως, αυτή η ανησυχία δεν θα πρέπει να εμποδίσει τη συνεννόηση, διότι μέσα από τη συνεννόηση θα λυθεί και η ανησυχία του κλάδου. Υπάρχει μια δυσπιστία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενός από τους εταίρους της. Και αυτό είναι προβληματικό. Θεωρώ λοιπόν ότι η έγκριση της συμφωνίας θα ήταν πολύ θετικό. Ναι, αλλά κύριε Σάντσο Πεσέδο, κοιτάστε εμεί εδώ να καλύπτουμε πράγματα τα οποία και δεν λειτουργούν και, και πραγματικά δηλαδή έχω φτάσει. έχω ξεπεράσει όλα μου τα όρια. Πραγματικά δηλαδή βγαίνω από τα ρούχα μου. Εμείς είμαστε εδώ σε επιτροπές, σε μικτές επιτροπές και δεν μας θέλουν στις μικτές επιτροπές ως παρατηρητές διότι, διότι, διότι, λείπει διαφάνεια. Εγώ δεν μπορώ δηλαδή να, να, να καταπίνω κάθε φορά ό,τι τρίχες μου λένε και δεν έρχεται εδώ κανένας υψηλόβαθμος υπάλληλο να μας τα πει. Και μου λέει εδώ η Κομισιόν ότι εγώ κοροϊδεύω τους βουλευτές. Ε, όχι δα. Εγώ τα σκέφτομαι αυτά τα οποία λέω και πληροφορούμε και δεν δουλεύω κανέναν και δεν λέω ψέματα σε κανέναν. Και πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί μου τα λέει η Κομισιόν αυτά. Εγώ μιλάω μια χαρά τα Ισπανικά και δεν καταλαβαίνω Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει κύριε Ραντούστ. Ε, συμφωνώ μαζί σας, είναι αξιοσημείωτα αυτά τα πράγματα, γιατί και εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να με ενημέρωσαν, ίσως στις διακοπές, δεν ξέρω, αλλά ξέρει τότε και η Κομισιόν πως λείπουμε, δεν μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας. Ε, δεν είχαμε λοιπόν πριν κάποια πληροφορία, από το ερώτημά μου προς την Κομισιόν είναι αν ε, μπορεί να μας ξαναστείλει αυτές τις πληροφορίες που υποτίθεται ότι λάβαμε για να δούμε και εμείς ε, πότε ε, υπήρχαν αυτές τις πληροφορίες. Συμφωνώ λοιπόν με αυτό το οποίο λέει η Πρόεδρος και δεν θα συμφωνήσω ε, με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Χωρίς να έχει αποφασίσει η ομάδα εργασίας μου, το κάνω εγώ μόνο μου, με δική μου ευθύνη. Αλλά έχω πάντα βεβαίως πρόβλημα όταν ή αυτοί οι οποίοι κάνουν ε, πολιτική, δηλαδή αφενός ε, οι Ισπανοί οι ψαράδες ε, και από την άλλη όσοι αλλιεύουν αυτά τα σκουμπριά και τα λοιπά ήδη αν δεν μπορούν να έρθουν σε μια συμφωνία και βλέπουμε εδώ πέρα μια συμφωνία η οποία δεν θα βοηθάει ούτε τους Ισπανούς, Ψαράδες, σε κανέναν άλλο και δεν ξέρω τελικά τι κάνουμε. Ας δούμε και στο παρελθόν τι είχε γίνει. Εγώ κατά κανόνα είμαι υπέρ της ε, πρόοδου και την ε, υποστηρίζω, αλλά αυτό εδώ πέρα πάρα πολύ δύσκολα. Προσωπικά εγώ δεν θα το υπερψηφίσω. Ευχαριστώ πολύ κυρία, κυρία Ανδρέας Μπαρέα. Κοιτάξτε, το θέμα είναι πολύ καυτό. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να το κρυώνουμε λίγο το πράγμα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να ξαναβρούμε την ψυχή όμως να οπισθοχωρήσουμε στις θέσεις μας. Υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές μεταξύ μας. Λοιπόν, εδώ ε, φαίνεται να υπάρχουν πληροφορίες που εδόθηκαν και υποσχέσεις οι οποίες δεν εκπληρώθηκαν. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έπρεπε να ξανακαλέσουμε την Κομισιόν εδώ με όλα μας τα ερωτήματα και με όλες μας τις απορίες και να ακούσουμε και τους αρμόδιους σε θέματα λίες και τους αρμόδιους για θέματα εμπορίου. Διότι εδώ έχουμε αντιφάσεις. Αναφέρθηκε η Πρόεδρος σαφέστατα στην έλλειψη συντονισμού μεταξύ των δύο γενικών διευθύνσεων. Το να ξαναδιαπραγματευτούμε τη συμφωνία μπορεί να είναι δύσκολο Αλλά τουλάχιστον μπορούμε να βάλουμε μία ρήτρα που θα μας βοηθούσε να λύσουμε το πρόβλημα. Αλλά πρώτα απ' όλα να ζητήσουμε από την Κομισιόν να μας δώσει καθαρότερες και περισσότερες εξηγήσεις από αυτές που δίνει. Ο κύριος Γκάλαχερ είπε και τώρα μιλάω ως κύριος Γκάλαχερ για να σας πω εγώ το Εμένα φέτος το καλοκαίρι που ήξερα δηλαδή πώς είχαν τα πράγματα, ούτε καν μου πέρασε από το νου να πάρω τηλέφωνο τον κύριο Γκάλαχερ και να του πω κύριε, κύριε Γκάλαχερ ε, να τον επηρεάσω οτιδήποτε και ο κύριος Γκάλαχερ μου τηλεφώνησε για να μου πει πόσο τσαντισμένος ήταν διορθώνεται μετά η πρόεδρος και λέει θυμωμένος Αυτά μου είπε λοιπόν. Εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Μπορούμε να υπερψηφίσουμε, να καταψηφίσουμε ή να καταθέσουμε τροπολογίες. Ο κύριος Αρσένης. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα περισσότερες ε, πληροφορίες. Νομίζω πως μια πιο ενημερωτική συνάντηση με την ε, Κομισιόν όπως αυτή την οποία πρότεινε η συνάδελφος, ε, θα μας βοηθούσε. Και συμφωνώ με αυτό το αίτημα. Bueno, de eh, quiero decir, como eh, el, eh, el 29... Στις 29 Σεπτεμβρίου είχαμε προβλέψει να ψηφίσουμε. Λοιπόν, μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε. Εμείς είχαμε πει ότι θα ψηφίζαμε είτε υπέρ είτε κατά. Η ψηφοφορία είναι το τελευταίο. Μπορούμε να το συζητήσουμε στις 29 και άμα δούμε ότι είμαστε έτοιμοι για να ψηφίσουμε, ε, τότε να ψηφίσουμε. Και όσο ενδιαφέρον και να είναι το θέμα, δηλαδή η χίλη και τα λοιπά, δεν μπορούμε να, να, να, να το κρατάμε εδώ για αιτίες. Τώρα η Κομισιόν το ξέρει πάρα πολύ καλά ότι εδώ εμείς είμαστε πολύ λογικοί σε αυτά που προτείνουμε. Απλώς η Κομισιόν τώρα έχει, ε, έχει ένα άχθος, έχει ένα πρόβλημα το οποίο θέλει να λύσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και κοιτάει να το ξεφορτωθεί. Είναι ένα πρόβλημα λοιπόν με τη Χιλή που πρέπει να το λύσουμε, διότι η Χιλή τι λέει ότι Λέ, η Χιλή λέει ορίστε αυτό είναι το πρόβλημα άμα σας αρέσει άμα δεν σας αρέσει. Και είναι αδιάλακτη η Χιλιανή και για τα θέματα αλλίας όπως και για τους ανθρακορίχους. Εγώ είπα ότι μέχρι μπορούμε να ψηφίσουμε ναι ή όχι, δεν είπαμε τροπολογίες, προθεσμία για τις τροπολογίες. Είπαμε να ψηφίσουμε ναι ή όχι στην πρόταση ψηφίσματος. 8. Πρόεδρε. Α, συγγνώμη, δεν σε είδα, δεν σε είδα, πραγματικά. Δεν σε είδα. Λοιπόν, ο κύριος Γκάλαχερ δεν είναι εδώ. Το θέμα της κυρίας Μπιλμπάο για τις αντσούγες και τα θέματα του κυρίου Γκάλαχερ τα είχαμε ήδη συζητήσει. Και μετά Είχαμε κάνει ένα γύρο ανατολιστικό για να δούμε τι θα κάνανε οι διάφοροι συντονιστές κτλ. Δεν ξέρω αν είχαμε, έχουν και τις πρώτες επαφές δηλαδή. Δεν είχαμε όμως άλλα νέα. Τώρα αυτό το οποίο είχαμε συμφωνήσει είναι αν θα συνεχίσαμε την ίδια πορεία ε, συζητώντας με την Κομισιόν ή αν θα ψηφίζαμε. Και θα πηγαίναμε και για λογαριασμό μας στην Ολομέλεια. Εδώ είχαν ακουστεί διάφορες γνώμες. Τώρα επειδή έχουμε εδώ την εισηγήτρια για τις αντσούγες, της δίνουμε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Λοιπόν, καλωσορίζω για τη νέα σχολική χρονιά, λέει η συγγήτρια όλους, ακόμη και τους διερμηνείς. Λοιπόν, στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Αλίας τον Ιούλιο είχαμε ένα πρόβλημα. Δεν θα σας κάνω καμία περίληψη για αυτό το σημείο αναλυτική, γιατί και εδώ υπάρχει έλλειψη διαφάνειας. Υπήρχε όμως ένα πρόβλημα σχετικά με τη νομική βάση που θα έπρεπε να εφαρμόσουμε, να εφαρμόσει το Συμβούλιο. Τώρα στην Επιτροπή Αλλιές είχαμε αποφασίσει, επειδή δεν είχε λάβει θέση το Συμβούλιο, να περιμένουμε το Σεπτέμβριο για να δούμε αν είμαστε σε θέσεις να συζητήσουμε ή να διαπραγματευτούμε με τη νέα Προεδρία το περιεχόμενο προσανατολισμού της Επιτροπής Ραλίας. Νομίζω ότι είναι βεβαιασμένη η κατάσταση σήμερα και το Συμβούλιο ήταν διακοπές και όλοι μας. Δύσκολο μου φαίνεται να έχουν καταλήξει σε κάτι, εκτός πια και αν σήμερα κάνουν καμία φοβερή αποκάλυψη που δεν πήραμε χαμπάρι κανένας. Ε, λέω λοιπόν να τα αφήσουμε το θέμα γιατί δεν ξέρουμε ποια είναι η θέση του Συμβουλίου για την νομική βάση και στη νέα κυκλική προεδρία αρμόδια για την αλία και αυτή δεν το είχε σαφές το πόσο θα αντιμετώπιζε το περιεχόμενο της προσανατολιστικής ψηφοφορίας της Επιτροπής Αγίας. Και αυτό που μας είπαν λοιπόν οι προεδρεύοντες ε, πριν από τις διακοπές ήταν ότι δεν το είχαν καθόλου με καθόλου καθαρό το θέμα. Θα έλεγα λοιπόν να το αναβάλουμε το θέμα για την επόμενη επιτροπή και να εξετάσουμε τα δύο θέματα εκ και τις εκθέσεις Γκάλαχερ όσο και τις αντσούγες. Κυρία Μπιλμπάου, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εμείς στην τελευταία συνεδρίαση αποφασίζαμε ότι δεν θα αποφασίζαμε προς την προηγούμενη συνεδρίαση γιατί θα το φέρναμε το θέμα σε αυτήν τη συνεδρίαση. Αυτό είναι καθαρότατο. Λοιπόν, ετέθη το θέμα στην ημερήσια διάταξη γιατί το είχαμε αποφασίσει στην προηγούμενη συνεδρίαση. Δεν έχω βέβαια κανένα πρόβλημα να αναβληθεί, εσείς θα το αποφασίσετε. και να βρούμε δηλαδή κάποια στιγμή και εδώ στην Επιτροπή μας μια λύση γιατί τελικά όμως αν το Συμβούλιο δεν αποφασίζει και εμείς δεν αποφασίζουμε κανένα θεσμικό όργανο δεν θα αποφασίσει. Τι να πω τώρα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με την πρώτη ανάγνωση, δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη λύση αν το Συμβούλιο δεν αποφασίσει. Αλλά εσείς οι σχεώδεις συγγητές να το λύσετε με τους συντηρηστές... και να μου κάνετε μία πρόταση για το πώς θα το λύσουμε. Πρέπει να βγούμε από αυτό το διέξοδο. Δεν μπορούμε εδώ δύο χρόνια να είμαστε ε, περιμένοντας να λάβουμε μια απόφαση γιατί το Συμβούλιο δεν αποφασίζει. Πρέπει να αποφασίσουμε. Και εμείς είμαστε υπεύθυνοι να αποφασίσουμε για τα διάφορα θέματα. Έχετε το λόγο κυρία Μπιλμπάου. Σύμφωνο απόλυτα μαζί σας. Η Επιτροπή γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι αυτό το θέμα Αυτό το θέμα με όλα του τα προβλήματα εξετάστηκε σύντομα, από μένα τουλάχιστον όσο εξαρτιότανε, γρήγορα. Απλώς αν καθυστερεί και αν τελματώνει το θέμα, τελματώνει λόγω του Συμβουλίου, για τη Ισπανική κυβέρνηση και η γαλλική κυβέρνηση ζήτησαν από το Συμβουλίο να παραλύσει το θέμα. Και μετά προέκυψε και το θέμα της νομικής βάσης, πράγμα το οποίο μας εξέπληξε γιατί κανένας μας δεν το είχε πάρει χαμπάρι. Και η Βελγική Προεδρία δεν ήξερε καθόλου εάν θα προχωρήσει, ήθελε να το προχωρήσει το θέμα. Απλώς και οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου που είναι παρόντες να μας πούνε μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτήν την προσωρινή ψηφοφορία, την προσανατολιστική ψηφοφορία που έγινε στην Επιτροπή μας. Να μας πούνε αν έχουν ξεκαθαρίσει κάτι για την νομική βάση. Εγώ είμαι έτοιμη να προχωρήσω σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Αλλά η Ισπανική και η Γαλλική κυβέρνηση αποφάσισαν να παραλύσει το θέμα. Λοιπόν μπορούμε να προχωρήσουμε άμεσα. Αν είναι δυνατόν να το ξεκαθαρίσουμε. Εγώ δεν θα ήμουν αντίθετη να συγκαλέσουμε μία συνεδρίαση αύριο και να το αποφασίσουμε και με τους σκεώδεις εισηγητές κλπ. Αλλά να ξέρετε ότι αν το θέμα έχει κολλήσει, αυτό είναι λόγω των εμποδίων της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Άντρεν Μπαρέα. Μας είπανε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα νομικής βάσης και η Κομισιόν δεν δεχόταν τους όρους μας και είχαμε ζητήσει να τοποθετηθεί και η Κομισιόν και πια φτάσαμε 30 Αυγούστου. Εγώ είχα προτείνει να έχουμε πρόταση από την Κομισιόν. Είμαστε στα τέλη Αυγούστου. Έχουμε λοιπόν εμείς το Σεπτέμβριο μπροστά μας, ας μας πούνε δηλαδή τι λένε για τη νομική βάση. για να μην έχουμε και ένα, θέμα, ένα πρόβλημα αρμοδιοτήτων. Αλλά να ξέρετε ότι το Συμβούλιο πραγματικά γυρνάει γύρω-γύρω. Μας ζαλίζει. Δεν Ζαλίζει την πέρβικα λέμε στα ισπανικά, στα ελληνικά αλήθεια πώς θα το λέγαμε λέει η πρόεδρος. Γυρίζει λοιπόν γύρω από το θέμα και μας ζαλίζει το Συμβούλιο και δεν μπορούμε να αποφασίσουμε. Φτάνουμε σε μία πρώτη ανάγνωση, ωραία, και ας έρθουν εδώ με την πρώτη ανάγνωση για να μας πούνε α, β, γ και άντε να αποφασίσουμε. Ή αλλιώ α τα αφήσουμε δηλαδή στι Ρωμαϊκέ καλένδε. Αλλά αυτό εμένα δεν μ' αρέσει γιατί εμένα μου αρέσει να αποφασίζω. Περιμένουμε λοιπόν το Συμβούλιο αλλά το Συμβούλιο δεν κάνει τίποτα ζαλίζει την περδικούλα μας. Ζητώ λοιπόν, μία προθε... δίνω μία προθεσμία σε εσά και τον κύριο Γκάλαχερ να ξεκινήσετε 15 μέρες μία διαβούλευση και να αποφασίσετε ποια διαδικασία θα ακολουθήσουμε. Διότι το Συμβούλιο μας ζαλίζει την περδικούλα. Άρα τι θα κάνουμε, Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου. Ζητώ λοιπόν σε 15 μέρες βρείτε τα με τον κύριο Γκάλαχερ και τους κοιόδης συζητητές και ελάτε να μου πείτε τι αποφασίστε. Η αντιπροσωπεία του Συμβουλίου είναι εδώ, να τους δώσω το λόγο, δεν πρόκειται να μου πει κουβέντα το Συμβούλιο. Θέλετε το λόγο Συμβούλιο. <coughs> Για να δούμε αν θα μας ξεκαθαρίσετε κάτι. Um, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν ε, είχα προβλέψει να επέμβω και νομίζω ότι έχετε δίκιο. Δεν θα πω και πολλά. Απλώς ε, η κυρία Μπιλπάου έχει δίκιο όταν λέει ότι φέτος το καλοκαίρι δεν έγινε μεγάλη πρόοδος, δεν είχαμε πολλές συνεδριάσεις, πιέζουμε και ίσως όλοι γνωρίζετε ποιο είναι το πρόβλημα και τι συζητάμε. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να επανέλθουμε σύντομα με μία τοποθέτηση του Συμβουλίου επί του θέματος, αλλά σήμερα δεν μπορώ να σας πω ότι έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Λοιπόν, πραγματικά επιβεβαιώνεται το όλο σε είπε. Εγώ βεβαίως δεν τα ρίχνω αυτά στην, ε, στη, στην καμπούρα της Βελγικής Προεδρίας. Αυτό το θέμα σέρνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ζητώ λοιπόν ε, οι δύο εισηγητές να συναντηθούν με αυτούς που πρέπει και να βρούμε ποια είναι η διαδικασία. Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, είμαι αρκετά ξεκουραστή μετά τις διακοπές. Λοιπόν, πάμε στα διάφορα και έχουμε το θέμα της κυρίας Ντόντ, διότι έθεσε το πρόβλημά της προηγουμένως, να τα ξαναπεί και να αποφασίσουμε σχετικά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Όλοι μάλλον στις τηλεοράσεις το καλοκαίρι είδαμε κάποια από τα θέματα που προέκυψαν σχετικά με σχετικά με το Σαβρίδι. Θα, δεν θα αναφέρω τώρα όλα αυτά τα ζητήματα, απλά θα σας πω τα σημαντικότερα σημεία της υπόθεσης. Την τελευταία δεκαετία ο κλάδος αυτός στην δυτικη Ευρώπη και στην Νορβηγία εργάστηκε για να διαχειριστεί τα αποθέματα τα δυτικά του Σαββριδιού αυτού έτσι ώστε διεθνώς να πιστοποιηθεί από το MSC ως αηφόρος ε, αλλήλια και αυτό ήταν υποδιαχείριση ε, μιας ε, συμφωνίας των κρατών αυτών που βρέχονταν από αυτή την θάλασσα και βεβαίως η ISIS θεώρησε πως υπήρχε μια προσέγγιση η οποία ήταν σύμφωνη με την αρχή της ε, προφύλαξης. Επειδή βεβαίως οι μη δεν ε, συμμετέχουν, δεν θα υπάρξει συνολική διαχείριση του αποθέματος αυτού το 2010. Γνωρίζουμε όλοι πως ε, κατέρευσαν οι διαπραγματεύσεις στο Λονδίνο τον Ιούνιο πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές και σε 7 Ιουλίου εγώ μαζί με άλλους Βρετανούς Ευρωβουλευτές και τους επικεφαλής του κλάδου από το Ηνωμένο Βασίλειο. Συναντηθήκαμε την κυρία Δαμανάκη για το θέμα αυτό. Εντυπωσιαστήκαμε από το πόσο στηρίζει την θέση μας. Αντιλαμβάνουμε ότι έκτατε η Επίτροπος συναντήθηκε και με τον Υπουργό Αλίας από τις νήσους ε, Φαρόες και απάντησαν με το να ανακοινώσουν μια δική τους ποσόστοση 85.000 τόνων. Εάν δούμε βεβαίω και τις μονομερείς ποσοστώσεις της Ισλανδίας, μιλάμε για ένα 35% του συνολικού επιτρεπόμενου αλλιεύματος για το Σαβρίδι, όπως έχουν συμφωνήσει τα κράτη αυτά, τα παράκτια. Το έχουμε συζητήσει αυτό επί μακρόν. Δεν έχει νόημα να το επαναλάβουμε το θέμα αυτό δηλαδή της Ισλανδίας και των ε, νήσων αυτών που μόνο μερός ανακοινώνουν τόσο υψηλές ε, ποσοστώσεις αναφέρουν ε, πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν αριθμοί σαβριδιού αν προηγουμένου τα ύδατά τους ως δικαιολογία. Γνωρίζουμε λοιπόν πως το σαβρίδι είναι ένα είδος μεταναστευτικό και αλλάζουν λοιπόν οι αριθμοί του. Οπότε προσωρινέ αυτές αλλαγέ δεν πρέπει να αποτελέσουν δικαιολογία για την υπεραλίευση. Η υπεραλίευση στην οποία οδηγούν βεβαίω αυτές οι αυξημένε ποσοστώσει και είναι κάτι το οποίο οι αλληλεί μας ε, που αλλιεύουν στην ανοιχτή θάλασσα προσπαθούν να αποφύγουν ε, τα τελευταία χρόνια. Η Νορβηγία αντέδρασε στις ανακοινώσεις αυτές με το να απαγορεύσει σε σκάφη από τις νήσους ε, Φαρόες ε, και Ισλανδία να εκφορτώνουν στις ηχθιόσκαλες τις δικές της και την ίδια πολιτική προτείνω να ακολουθήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και πριν από λίγες εβδομάδες και το ίδιο προτείνω και σήμερα. Εάν δεν υπάρξει τέτοια πολιτική πρέπει να συγχαρώ τους ε, Σκοτσέζους ψαράδες που εμπόδισαν την εκφόρτωση από ένα σκάφος με σημαία νήσων φαρών πριν από λίγες εβδομάδες στο Πίτερχετ. Για εμάς λοιπόν όλα αυτά θυμίζουν μια υπόθεση πριν από λίγα χρόνια που είχε ως αποτέλεσμα να ανταμυφθεί η Ισλανδία με μια πάρα πολύ υψηλή ποσόστοση για ένα άλλο είδος το οποίο τώρα είναι στα όρια τη εξαφάνισης. Με συγχωρείτε λέει η πρόεδρος. Ε, που σα διακόπτω, αλλά κοιτάστε έχουμε καταλή... πρέπει να διακόψω τη συνεδρίαση σε 3-4 λεπτά, διότι έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Να είστε σύντομοι λοιπόν. Ναι, σχεδόν τελείωσα. Να υπενθυμίσω στην Επιτροπή πως η Ισλανδία αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει και διαπραγματεύσει ένταξη στην Ένωση να ζητήσω επίσης η Επιτροπή μας να καταγράψει την στήριξή μας για την Επίτροπο Δαμανάκη και την στεναρή της στάση και καλούμε Κομισιόν και κράτη-μέλη να σκεφτούν να αναλάβουν μέτρα, τα κατάλληλα μέτρα και μάλιστα κυρώσεις εις βάρος των δύο αυτών χωρών. Όπω έκανε και η Νορβηγία. Επίση, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στην Ισλανδία πω εδώ πέρα κινδυνεύουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσει του με αυτή την κατάφορη αδιαφορία ε, διεθνών, ε, για τις διεθνείς συμφωνίες. Επίσης, υπάρχει την ερχόμενη εβδομάδα διάσκεψη της νησφαρόες για αυτό ακριβώς το ζήτημα και μάλιστα ηρωνικά αφορά τις πτυχές διαχείρισης αυτού του συγκεκριμένου αλλιεύματος. Θα ήθελα λοιπόν η Κομισιόν να αποστείλει μια μικρή αντιπροσωπεία στη διάσκεψη αυτή. Αντιλαμβάνομαι πως ε, η Κομισιόν και κάποια κράτη-μέλη επίσης θα εκπροσωπηθούν. Ε, και σας ευχαριστώ που μας επιτρέψατε να θέσουμε αυτό το θέμα στην Επιτροπή είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον κλάδο συνολικά. Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο μιλάμε για 150 εκατομμύρια λίρες ε, το χρόνο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Τόμσον, αλλά θέλω να τον ρωτήσω. Αυτή η πρόταση της κυρίας Ντότς και Στίβανσον θα μπορούσε ας πούμε ένας αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας να πάει ως μέλος της κοινοτικής αντιπροσωπείας σε αυτή τη διάσκεψη που θα γίνει στις ε, Φερόε Δεν ξέρω, να δούμε τι θα πει ο κύριος Τόμψον. Εγώ θα έλεγα ο κύριος ε, Στίβενσον που είναι και πρώτος αντιπρόεδρος και σκοτσέζος να μας εκπροσωπήσει σε αυτή τη συνεδρίαση στις αρχές Σεπτεμβρίου. Συμφωνείτε? Ωραία. Ο κύριος Τόμψον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως πολύ σωστά τονίσατε σήμερα, πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτή την εποχή σχετικά με την διαχείριση του σαφριδιού στο Βόρειο Ατλαντικό. Και όπως πολύ σωστά είπατε, η Επίτροπος ε, έχει αναλάβει μία πολύ στεναρή ε, θέση σχετικά με την αλληλεία στο Βόρειο Ατλαντικό και πιστεύουμε ότι τις τελευταίες εβδομάδες η στάση ε, των ε, νήσων Φαρό δεν ήταν πολύ σοβαρή. Η Επίτροπος λοιπόν έχει απευθύνει μία ε, προσωπική επιστολή εις τον υπεύθυνο Υπουργό Αλληλείας σχετικά με τα τεκτενόμενα και είχαμε αρχές Αυγούστου με τους ενδιαφερομένους και τη βιομηχανία για τις διαμαρτυρίες που θα απευθυνθούν προς τις νήσους Φαρό και ίσως και την Ισλανδία. Προς το παρόν όμως ιδίως στις νήσους Φαρό. Και ε, είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε. Τίποτα δεν αποκλείεται αυτή τη στιγμή κυρία Πρόεδρε. Ε, ε, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το επόμενο βήμα θα είναι να έχουμε μια συνάντηση με τις νήσους Φαρό και θα προσπαθήσουμε στα μέσα αυτής της εβδομάδας ή την επόμενη εβδομάδα να την οργανώσουμε και ελπίζουμε ότι ο εκπρόσωπος των νήσων Φαρό θα είναι στην συνεδρίαση που ανέφερε η προλαλήσασα στις αρχές της επομένης εβδομάδας, οπότε φαντάζομαι ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα μπορέσουμε να τον έχουμε συναντήσει. Όσον αφορά τους εκπροσώπους αυτής της Επιτροπής θα πρέπει να επανέλθω αφού το συζητήσω με τους υπευθύνους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, αλλά νομίζω ότι εδώ μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για το θέμα. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να εργάζεται επί του συγκεκριμένου θέματος πολύ θετικά διότι υπάρχει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι ικανοποιητικό για όλους ενδιαφερομένους μόνο, όχι μόνο την κοινότητα αλλά την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Φαρό και την Ισλανδία. Θα ήθελα λοιπόν να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι ε, ε, ικανοποιητικό για την βιομηχανία αλίας ανοιχτής θαλάσσης ε, και να μπορέσουν να συμμετάσχουν και μέλη της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μας είναι δυνατόν να λυθεί το θέμα το ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ κύριε Τόμψον, ευχαριστώ και τους ε, διερμηνείς που μας άφησαν πέντε λεπτά παραπάνω. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε ο κύριος ε, Στίβενσον να μας εκπροσωπήσει σε αυτή τη διάσκεψη για να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Λοιπόν, 29 Σεπτεμβρίου επόμενη συνεδρία, πέρας τη συνεδρία.